με τους μαλαισινούς φίλους. Ελπίζουμε η επίσκεψή σας να είναι καρποφόρα και ενδιαφέρουσα. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μπροκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, Αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως είναι ένα κλασικό παράδειγμα αντιευρωπαϊσμού που δεν κατανοεί το περιεχόμενο της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αλλά θα ήθελα τώρα να σταθώ στη σημερινή συζήτηση. Η, Ευρω... η Σουηδική Προεδρία με μεγάλη ικανότητα και επιδεξιότητα και εμπιστοσύνη μπόρεσε να εξασφαλίσει και την κύρωση της ε, Συνθήκε της Λισαβόνας. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί χρειάστηκαν εννέα χρόνια για να έλθει το πλοίο επιτέλους σε ασφαλή λιμένα. Επιτέλους λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε στην πράξη τις ρήτρε της ε, τη της Λισαβόνας χωρίς αυτό να προσκρούει σε κάποιο νομικό κόλλημα. Πρέπει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λοιπόν να έχει μια πραγματική νομιμοποίηση και να εκλέγεται όχι μονάχα από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων, αλλά εν καιρό από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει μια πλήρη νομιμοποίηση. Επίσης, είναι απαραίτητο να τονίσω πόσο σημαντικά ήταν, όπως είπε ο Ζαρμονέ, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο ύπατος εκπρόσωπος να αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Δεκεμβρίου ως ε, ύπατος εκπρόσωπος και μετά να επανέλθει ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Όχι, μόνο με την πλήρη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δυνατόν να αναλάβει τα καθήκοντά του και δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρεξήγηση σε σχέση με το θέμα αυτό και σας τονίζω ότι και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσει τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε αυτό να είναι μια ευκαιρία για να γίνει μια εγκρυπτό διακυβερνητικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Και εμείς δεν θα δεχτούμε οτιδήποτε το οποίο θα διαταράξει την ισορροπία εξουσιών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο Ενάμιση λεπτό, λεπτό Άντριαν Σεβερίν. Κυρίες και κύριοι, η θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα είναι ένα ιστορικό συμβάν, ένα ιστορικό γεγονό. Θα πρέπει να χειροκροτήσουμε, να εκφράσουμε την, ευγα... την ευαρέσκειά μας και θα πρέπει να συγχαρούμε φυσικά και τη Σουηδική Προεδρία για την προσπάθεια την οποία έκαναν για να πετύχουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μια συνθήκη παρόλα αυτά από μόνη της δεν αρκεί, αφού αυτής δεν αρκεί και η τέλεια συνθήκη από μόνη της δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε εμπνευσμένου ηγέτε για να την εφαρμόσουν. Στην περίπτωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γιατί η συνθήκη αυτή είναι καρπό συστηματικών συζητήσεων, μακρόχρονων συμβιβασμών και είναι αναπόφευκτο η συνθήκη αυτή περιλαμβάνει πολλά διφορούμενα στοιχεία και ίσως και πολλά κενά. Γι' αυτό ακριβώς οι μελλοντικοί πολιτικοί θα πρέπει να διευκρινίσουν τα κενά αυτά, να μπορέσουν να μορφοποιήσουν τα όργανα και να δώσουν τις σωστές ερμηνείες σε όλες τις ρήτρες της συνθήκης, να ορίσουν τους ρόλους και τις αποστολές. Ακριβώς η επόμενη εντολή όλων αυτών των προσώπων που αναζητούμε θα είναι κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την συγκεκριμένη θεσμική αρχιτεκτονική. Για να είναι βιώσιμη η αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να είναι σύνθεση όλων των πολιτικών εμπειριών, των πολιτικών κληρονομιών αν θέλετε ε, και των πολιτικών πολιτισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ήπατος για τα εξωτερικά θέματα θα πρέπει να εκφράζουν όλες τις πολιτικές επαισθησίες, όλες τις γεωπολιτικές περιοχές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα το πετύχουμε και ελπίζω επίσης ότι ακόμα και όταν το πετύχουμε αυτό θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της θεσμικής μας αρχιτεκτονικής, την αποτελεσματικότητα των οργάνων και την αξιοπιστία της Ένωσης στα μάτια των πολιτών μας. Η κυρία Ανελή Γέτενμάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά εξαίρεση, θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω τον τύπο. Θέλουμε να υπάρχει πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλιώς οι πολίτες δεν θα συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς συζητείτε το θέμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτές τις τρεις θέσεις για τις δύο θέσεις για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον είπα το εκπρόσωπο. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα υποψηφίων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι δημοκρατικές εκλογές. Ε, είχαμε εκπροσώπους του, της Βουλής ε, της ε, Τουρκίας παρόντες όταν συζητούσαμε το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας και μας ρώτησαν τότε πώς ακριβώς θα διοργανώσετε τις εκλογές, πώς θα επιλέξετε τους υποψηφίους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Άσλι Φόξ. Ο κυρίος Φόξ, συγγνώμη, πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις άτυπες συζητήσεις που έγιναν πέρσι στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο για την επιλογή φυσικά του επόμενου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το ρόλο που θα διαδραματίσει πιστεύω ότι ο πρόεδρος πρέπει να υπηρετεί το Συμβούλιο, να είναι ένας ε, πρόεδρος και έχει ένα ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος. Είναι σημαντικό ο πρόεδρος ε, να, ε, να χαίρει της εμπιστοσύνης και των πολιτών και του σώματος και να επιλεγεί από αυτό. Οπότε... Μόνο ο Τόνι Μπλερ θα ήταν καλός υποψήφιος για αυτή τη δουλειά και όπως είπε η κυρία Μέρκελ, φοβάμαι μην χρειαστεί ε, να ακούω για πέντε χρόνια τον κύριο Πλάσο όσο περνάει το αυτοκινητοπομπή του. Ε, και το θέμα της εμπιστοσύνης έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, δυστυχώς πολλές φορές ε, ο κύριος ε, Μπλαερά έχει δείξει πόσο αναξιόπιστος είναι. Δεν μπορεί να κατέχει δημόσιο αξίωμα και σας απευθύνω έκκληση να μην τον διορίσετε. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Ο κύριος Μπάστιαν Μπέλντερ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα με ενδιαφέρον ε, την ε, παρουσίαση, το έγγραφο της Σουηδικής Προεδρίας για την ε, εξωτερική δράση και είναι καλό που η Σουηδική Προεδρία έχει προβλέψει περισσότερο χρόνο για την επιλογή του υποψηφίου για τη θέση του υπατέκ προσώπου. Δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να, ε, καλύψουν αυτή τη θέση. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ γιατί το διακύβευμα είναι η διαθεσμική εσωτερική ισορροπία. Πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου και η εξωτερική δράση είναι η εξωτερική πολιτική, είναι θέμα κατά βάση εθνικής αρμοδιότητας. και παρά τις καλές προθέσεις ε, νομίζω ότι δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας. Ε, ο κύριος Φίλιπ Κλέης τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο έχει λάβει η χώρα. Εμείς, παραγματικά στο Βέλγιο, αντιμετωπίζουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Φαν Ρομπέι και βλέπουμε ότι απλώς τον προωθούν γιατί είναι πολύ καλός στο να βρίσκει συμβαστικές λύσεις και δεν δημιουργεί καμία ε, εχθρότητα. Κάποιος ο οποίος μπορεί να διοικεί το Βέλιο μπορεί να διοικεί ίσως και την Ευρώπη αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Ευρώπη χρειάζεται κάτι περισσότερο. Ο κύριος Φαν Ρόμπεϊ δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν επιτυχής σαν πρωθυπουργός. Το Βέλιο ουσιαστικά είναι μια κυβέρνητη χώρα και ο κύριος Φαν Ρόμπεϊ ουσιαστικά μονάχα μπόρεσε να διεκπαιρεώσει τις τρέχουσες υποθέσεις και τίποτα περισσότερο. Εμεί χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα είναι πιο ισχυρός μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο οποίος θα μπορέσει να υποστηρίξει όλα αυτά τα προβλήματα που, που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Κλέους. Ο κύριος Ότμαρ Κάρας. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από 20 χρόνια η βία διαίρεση της Ευρώπης σε μια περιοχή ελευθερίας και σε μια περιοχή δικτατορίας κατελήθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πολιτικό εγχείρημα το οποίο εξασφάλισε την επανένωση της Ευρωπαϊκής Υπήρου και το έκανε πραγματικότητα. Είναι αυτό το πολιτικό εγχείρημα η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση η οποία έχει σαν στόχο να γίνει μια ευρεία ζώνη δημοκρατίας, σταθερότητος, ελευθερίας και ευμάρειας μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια κοινότητα αξιών και μια κοινότητα στόχων η οποία θα διατηρηθεί. Πρέπει όλοι λοιπόν να συμβάλλουμε ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό. Χρειάζεται μια στεναρότητα και μια αποφασιστικότητα ώστε να μην ξαναυπάρξουν ποτέ πια τύχη μεταξύ τα οποία να χωρίζουν τους λαούς της Υπήρου μας. Και τονίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική προώθηση στην Ευρώπη μετά από την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί αυτή η συνθήκη δίνει στους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ο εκπρόσωπος μιας ολόκληρης υπήρου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία, πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη πολιτική θέληση για να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε την πρόεδρο αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό σημαίνει πολιτική θέληση. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια να λειτουργούμε με βάση τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Οποιαδήποτε αυτό εξαίρεση, οποιοδήποτε opt-out αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση στην Ευρώπη θα μπορέσει να ξεπεραστεί μονάχα όταν υπάρχει ανάπτυξη με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και χωρίς συμφωνίες οι οποίες αφορούν χρηματοδότηση τραπεζών με τεράστια ποσά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, το οποίο σημαίνει ότι ψάχνουμε πάντα για την καλύτερη λύση και όχι την πιο απλή. Οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει για, τα, για τις προσωπικότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μου δημιουργούν το φόβο ότι δεν ψάχνουμε για ευρωπαϊκές λύσεις, δεν ψάχνουμε για τους καλύτερους, αλλά για μια συμφωνία μονάχα πολιτικών κομμάτων. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που τροχοπέδησε την επίτευξη της κύρωση Συμφωνίας Λισαβόνα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Κάρας. Λόπες ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αντίστοιχες πτυχές των ε, συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την οπτική γωνία της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός χώρου δικαιοσύνης και ελευθερίας και εσωτερικών για τα θέματα μετανάστευση. Εγώ χαίρομαι για το γεγονό ότι εδόθη μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό στα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι στο μέλλον η πολιτική μετανάστευση θα είναι μια κοινοτική πολιτική και η Ισπανική Προεδρία έχει σαν πρόθεση να εμπλέξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πολιτική. Συγχρόνω, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και την αλληλεγγύη ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ ε, <clears throat> και λυπάμαι που δεν θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι πραγματικά υποχρεωτική αλληλεγγύη ιδίως στις χρηματικέ της πτυχέ. Πιστεύω ότι η διεύρυνση του χώρου συναπόφασης στα εσωτερικά και τα θέματα δικαιοσύνης είναι ένα σημαντικό βήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένουν πολλά από μας οι Ευρωπαίοι πολίτες και γι' αυτό είναι σημαντικό οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου να εδραιώσουν αυτό το χώρο εσωτερικών και δικαιοσύνη ως ένα μεγάλο χώρο κοινοτικού χαρακτήρα ευρωπαϊκό με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοχόλμης στον οποίο έχει ήδη συμβάλει η Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών με την έκθεση που θα εγκριθεί αυτή τη βδομάδα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά σεβαστήσατε το χρόνο τον οποίο είχατε στη διάθεσή σας. Ένα λεπτό κύριος Νταφ. Πρόεδρε, είναι καταπληκτικό που μπορούμε να κλείσουμε αυτό το, το τελευταίο κεφάλαιο του μυθιστορήματος της συνθήκης της Λισαβόνας. παρατείναμε το φτωχό προηγούμενο της Βρετανικής εθιμοτυπίας, αν θέλετε, δηλαδή τα όσα ε, έγιναν με τη χάρτα. Ε, και ως, ε, όπως συνηθίζουν θέλουν να έχουν μια ρήτρα opt-out από την συνθήκη. μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι ε, η Χαρτά Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ε, θα συνεχίσει να είναι δεσμευτική παρά τα όσα έκανε ο Τσέχος πρόεδρος που κάθεται και οι Τσέχοι γενικότερα που κάθονται στο κάστρο τους οχυρωμένοι. θέλουν να αποφύγουν το να μπορούν οι πολίτες να επικαλούνται τη χάρτα σε δίκες, σε δικαστικές διαφορές εθνικές. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πιωτρόφσκι. Κυρίες και κύριοι, Κυρίες και κύριοι, παρόλες τις διακηρύξεις για τον τρόπο καλύτερης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ουσία η συνθήκη αυτή είναι το κουτί της Πανδώρας τίποτα δεν διευκρινίζεται, οι ερμηνείες διαφέρουν και υπάρχουν ήδη διαιρέσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες. Κανένας δεν γνωρίζει το τι ακριβώς θα κάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει δημοκρατικός ουσιαστικός έλεγχος και το μόνο το οποίο θα κάνει είναι ίσως ε, κάποια πράγματα που έκανε στο παρελθόν τελετουργικά περισσότερο και ανάλογα με τον χαρακτήρα του προσώπου που θα καταλάβει τη θέση το για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι, περισσότερες, οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρωτώνται. Οδεύουμε προς ένα ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό υπερκράτος εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Ε, τι θα πρέπει να κάνει ένας Ευρωπαίος Πρόεδρος από το να επανέλθει στην αντιδημοκρατική πολιτική που ακολουθούσε στο παρελθόν η Ευρώπη. Ο Μάουρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη Σουηδική Προεδρία για τα κομβικά σημεία επιτυχίας τα οποία μας παρουσίασε αυτό το εξάμεινο. Θα ήθελα να σας κάνω και ένα δώρο, ένα, μια λευκή κόλλα χαρτί μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σαν μέσο για να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που παραμένουν ακόμα για τον σωστό εντοπισμό των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου του Συμβουλίου και του υπάτου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Να προσπαθήσετε να πείσετε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να γράψουν στο χαρτί αυτό όχι τα ονόματα που ακούμε δεξιά και αριστερά, αλλά τις ιδέες τις οποίες έχουν για την εξωτερική μας πολιτική. Αν το πετύχετε αυτό θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό προς τα εμπρός βήμα. Αν μας διευκρινίσουν ακριβώς το τι περιμένουν από μας, το τι περιμένουν από αυτούς, τότε θα είναι εύκολο να προσπαθήσουμε να ορίσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα και ονόματα. Αυτή είναι η πραγματική διαφάνεια την οποία απαιτούμε όλοι σήμερα. Θα πρέπει να δούμε τι ιδέα έχει ο κάθε αρχηγός κράτους για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να επιλεγούν πρόσωπα τα οποία να προσωποποιούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην διεθνή σκηνή για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τα ιδανικά των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικό ενωτικό στοιχείο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα μονολυθικό μπλοκ. Είναι καρπός δράσεων συγκεκριμένων προσωπικότητων και καλείται να ανανεώνεται συνεχώς. Η Ευρώπη θα πρέπει φυσικά να εκκινήσει εκ νέου στις αξίες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε, να χρησιμοποιήσει τις επιτυχίες της και με μια σωστή δόση ρεαλισμού όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο Για 1,5 λεπτό τον λόγο έχει ο κύριος Άσολη. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σουηδική Προεδρία για την προσπάθεια την οποία έκανε και για τις προσπάθειες για την τελική επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Το είχαμε ανάγκη αυτό. Έχουμε ανάγκη τη νέα συνθήκη γιατί μας δίνει επιπλέον την δυνατότητα να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες και αυτού εδώ του Κοινοβουλίου και έχουμε και δύο νέα πρόσωπα θα έλεγα τα οποία θα αντιπροσωπεύουν μια κάποια σύνθεση πολιτική και θεσμική. Γι' αυτό ακριβώς ευχόμεθα το Συμβούλιο εν την πλήρη αυτού σοφία να ερμηνεύσει τις, τα αιτήματα των μεγάλων πολιτικών οικογενειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε στα πλαίσια της επόμενης συνάντησής του να ορίσει με αποφασιστικότητα και αξιοπιστία τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να αναλάβουν ε, τις νέες θέσεις οι οποίες προβλέπονται από τη συνθήκη. Τι έχουμε ανάγκη λοιπόν. Έχουμε ανάγκη από με έναν πρόεδρο του Συμβουλίου που να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συνέχεια στην πολιτική μας. Έχουμε ανάγκη από έναν εκπρόσωπο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής που να μπορεί να χειριστεί τα προβλήματα που δημιουργεί μια διεθνής πολι- σκηνή πλέον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε και την κυβερνητική διάσταση και την κοινοτική διάσταση. Έχουμε ανάγκη επίσης και από ένα σύνολο επιτρόπων ισχυρό, ισορροπημένο και πολιτικά και σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και φυσικά εθνικά. Και είναι σημαντικό που κάτι τέτοιο συμβαίνει 20 χρόνια μετά από την πτώση του τείχους που διέρεσε την Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία θα πετύχουμε τώρα θα δώσουν νέες ελπίδες στους λαούς της Ευρώπης για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, για μια Ευρώπη δικαιοσύνης. Ευχαριστώ κύριε σας όλοι για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λουί Μισελ. Πρόεδρε, Προεδρεύουσα στο Συμβούλιο, θα αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Σουηδική Προεδρία για την πραγματικά αξιόλογη εργασία. Θα ήθελα επίσης ε, μέσω της κυρίας Μάλμστρομ να απευθυνθώ στον κύριο Μπαρόζο. Είμαι σίγουρος ότι θα μεταφέρει τα σχόλιά μου το ίδιο ε, και ε, για την παρέμβαση του κυρίου Φερχόφστατ. Θέλουμε να εξασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας του και θέλουμε με τόλμη να εφαρμόσει την κοινοτική μέθοδο. Αν αυτή την επιτροπή θέλουμε και από ό,τι κατάλαβα από την παρέμβασή του αυτό επιθυμεί ο κύριος Μπαρόζο, πρέπει να διαρθρώσει τη δράση του χρησιμοποιώντας την ομαδοποίηση των κατηγοριών σε πυλώνες και κάθε πυλώνας ε, θα υπόκειται στην αρμοδιότητα ενός αντιπροέδρου που θα έχει την, ε, όχι μόνο την αρμοδιότητα αλλά και την εξουσία να εξασφαλίσει την συνοχή όλων των πολιτικών που υπάγονται στον πυλώνα. Το κατακαιρματισμό που ισχύει τώρα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξέρω τι λέω γιατί υπηρέτησα πέντε χρόνια ως Επίτροπος. Αυτός ο κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων ε, υπονομεύει την κοινοτική μέθοδο και το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, και πλήττει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα το πείτε στον κύριο Μπαρόζο, ελπίζω και είναι δύσκολο φυσικά να ξανασχεδιάσουμε τις αρμοδιότητες ε, που έχουμε ε, κληρονομήσει από το παρελθόν λόγω κάποιων κυροσκοπικών μεθοδεύσεων, αλλά δεν πιστεύω ότι ο τωρινός πρόεδρος δεν θα αναγνωρίσει ότι χρειάζεται νέα φιλοδοξία για την νέα Επιτροπή. Ευχαριστώ τον κύριο κύριο Μισελ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Μπαρινιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Χάρη στην επιμονή της Σουηδικής Προεδρίας που θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, επικυρώθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά δεν είναι ένα σχέδιο, είναι ένα εργαλείο, ένα κουτί με εργαλεία που ε, υπηρετεί τους ε, πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπαλλήλους, όλα τα θεσμικά όργανα, λοιπόν, και όλοι οι θύνοντες πρέπει και εμείς εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τρόπο αυτά τα εργαλεία μετά από αυτήν την παρατεταμένη μεταβατική περίοδο. Εμεί είμαστε σε θέση για να αντιμετωπίσουμε τρει βασικέ προκλήσει και αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι από αυτό εξαρτάται όχι μόνο η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπω είπε και ο κύριο Βακλαβ εξαρτάται από αυτό η κυριαρχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η βασική ε, πρόκληση είναι να ε, αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν υπάρχουν ε, στοιχεία στις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ ε, για τα θέματα κυριαρχίας, θέματα διαφάνειας, θέματα ρύθμισης των ε, διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και εμείς από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, από την συμφιλίωση της αγοράς με το κοινωνικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως ανέφερε εξάλλου και ο Μπαρόζο. Δεύτερη πρόκληση, η πράσινη ανάπτυξη. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κιώτο έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο και πρέπει να τον διατηρήσουμε μεριμνώντας ώστε οι εταίροι μας, οι υπόλοιπε περιοχές του κόσμου να έχουν μια αντίστοιχη στάση. Τρίτη πρόκληση, ε, είναι δικό μας καθήκον να είμαστε στην ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτών που θα αποφασίσουν για την τάξη ή για την αταξία που θα επικρατήσουν στον κόσμο τα επόμενα 20 χρόνια. Εύκολο δεν είναι. Ε, Εκτό αν δεχτούμε, που εγώ δεν το δέχομαι, να δεχόμαστε την επιρροή άλλων χωρών. Ε, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον μελλοντικό ύπατο εκπρόσωπο ε, που θα ηγηθεί μια ενιαία δομή αρμόδια για την εξωτερική δράση. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί έχουν προσδοκίε οι Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένουμε την απόφασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό στην κυρία Κόγκ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας μιλήσω εδώ για την ε, έκθεση για τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά για τις οικονομικές επιπτώσεις του Συμβουλίου του των αποφάσεων του Συμβουλίου. Καταρχήν πρέπει να σας πω πώς εμφανίζεται η κατάσταση σε αυτό το έγγραφο. Αλλά πιστεύω ότι πλέον οι άνθρωποι δεν έχουν δυνάμεις, οι επιχειρήσεις ε, δεν έχουν πόρους και δεν έχουν δυνατότητα να λάβουν πιστώσεις. Και ε, χαίρομαι που όλα αυτά τα προβλήματα αντικατοπτρίζονται στο έγγραφο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η οικονομική ανάκαμψη δεν είναι ε, παρκής και η Ευρώπη είναι πιο ασθενής ε, τώρα. Η Ευρώπη αρχίζει να ενισχύεται αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες και να δημιουργήσουμε απασχόληση και να ε, καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εάν δεν κάνουμε όλα αυτά, δεν επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους, δεν θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει λοιπόν τα συστήματα αυτά να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά και όσον αφορά ε, την ε, κοινωνική Ευρώπη και όλα τα κεκτημένα, στα πλαίσια της οικονομικής Ευρώπης. Ε, αυτή είναι η εργασία μας και η ε, ευθύνη μας. Η κυρία Εκ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πολιτική και η ψυχολογία ε, προχωρούν από κοινού και αυτή τη στιγμή πολλοί προσπαθούν να μειώσουν τον απόϊχο ε, της ε, διασκέψεως της Κοπενχάγης σε λίγο καιρό και το αντιλαμβάνομαι διότι πολλές φορές έχουμε καταστρέψει τους, ε, κλιματικούς στόχους. Ε, δεν πρέπει λοιπόν και τώρα να ε, τους θάψουμε. Θα πρέπει γι' αυτό η Σουηδική Προεδρία να προχωρήσει αυτή την προσπάθεια την επικοδομητική διότι εάν δεν έχουμε μία δεσμευτική συμφωνία στην Κοπεχάγη δεν θα επιτύχουμε τους στόχους και ο βασικός στόχος είναι ο δευ... Ε, του δευτέρου βαθμού και γι' αυτό πρέπει να τον υλοποιήσουμε. Υπάρχουν δύο ομάδες ατόμων, αυτοί οι οποίοι ε, προχωρούν και αυτοί που απλώς κατακρίνουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σημειολόγησα αυτά ακριβώς που είπε η Προεδρία για την οικονομική κρίση αλλά είναι φανερό ότι εκτός μιας χώρας όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σύμφωνο σταθερότητας. η οικονομική κρίση άλλωστε τελικά δεν πρέπει να αποβεί σε κρίση αρχών και αξιών. στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής η προεδρία έπραξε πολύ σωστά. σημασία έχει όμως να πιέσει όχι μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και τις Ηνωμένε Πολιτείε, για να αλλάξει κατάσταση να αναλάβει τις πραγματικές πρωτοβουλίες στην κοπενχάγη. Στο τρίτο ζήτημα στη συνθήκη της Λισαβόνα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε ευτυχείς. Εννέα χρόνια μετά την κρίση που υπήρξε στη συνθήκη της Νίκαιας και την αδυναμία να απαντήσουν στο θεσμικό ζήτημα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνθήκη που αρκετοί μας ταλαιπώρησαν για να υπογράψουν. Σημασία δεν έχει μόνο ο θεσμός και η συνθήκη. Σημασία έχουν και τα πρόσωπα που την εφαρμόζουν. Και υπ' αυτή την έννοια η Προεδρία έχει ευθύνη και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής επιτροπής ώστε τα πρόσωπα που θα αναλάβουν κυρίως ο υπουργός εξωτερικών να εκφράζει το σύνολο των συμφερόντων των καλώς νοουμένων της ένωσης και από την άλλη πλευρά ε, στο επίπεδο του συμβουλίου τα περί του συμβουλίου είναι ζητήματα που πολλοί από εμά ε, δεν τα θέλαμε. εγώ προσωπικά ήμουν μέλος της ευρωπαϊκής συνέλευσης πολλοί από εμά δεν θέλαμε να υπάρχει πρόεδρο του συμβουλίου θέλαμε ο ρόλο αυτό να αναλυφθεί από τον πρόεδρο τη Επιτροπή και είχε συμβεί και στο παρελθόν διότι στην ουσία και ο ρόλο του προέδρου τη επιτροπής είναι να συντονίζει το συμβούλιο και να αποφεύγει τι περιπέτειες των συγκρούσεων. ευχόμεθα και η προεδρία της ευρωπαϊκής επιτροπής αλλά κυρίως η προεδρία του συμβουλίου να δώσει τις κατάλληλες συστάσεις στα κράτη μέλη ώστε ο τρόπος που θα λειτουργήσουν και τα δύο όργανα να είναι τέτοιος που να μην αφίσταται τη κοινοτική μεθόδου εργασίας και ενό καλού παρελθόντος που έχουμε στην ευρώπη που μας εξασφάλισε τόσα πολλά χρόνια ευημερία. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Ραμόν Ορέγγι. Έχει το λόγο ο κύριο Ραμόν Ορέγγι. Για μισή λεπτό. Πρόεδρε, Θέλω να πω ότι το πρόβλημα σχετικά με την Τσεχία, ή μάλλον η λύση του, μπορεί να μην ήταν τέλεια, αλλά ήταν η καλύτερη δυνατόν. Ήταν η καλύτερη δυνατόν για να μην έχουμε πιο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε νέους επίτροπους, νέα επιτροπή δηλαδή φέτος, έχουμε νέο ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέο νομικό καθεστώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρονιά αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική με το νέο νομικό της πρόσωπο. Δεν αποτελεί πια ε, μια συσσόρευση κρατών, αλλά αποτελεί μια νέα οντότητα. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε τη βούλησή μας να προχωρήσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τις ε, δυσκολίες αυτές των ρευμάτων εθνικισμού που μας εμποδίζουν να πάμε προς τα μπρος. Για σκεφτείτε, πριν από 10 χρόνια Πώς φανταζόμασταν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα πετυχαίναμε το ευρώ πριν από 10 χρόνια αν δεν είχαμε παραιτηθεί ο καθένα μας από την ε, πεσέτα, το φράγκο του κλπ. Δύο πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ότι η κατάσταση πήγε. Το Σώμα των Επιτρόπων το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο πρέπει να εγκριθεί. Είναι πολύ σημαντικό η επόμενη Προεδρία τον ε, Ιανουάριο να ξεκινήσει με ένα νέο σώμα επιτρόπων, που να το έχουμε ήδη από τα τέλη αυτής της χρονιάς. Και από εκεί και πέρα, λέμε βούληση πρέπει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βούληση για τι πράγμα. Για να ληφθούν οι μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι δυνατή και ενωμένη για να προχωρήσει με το δικό της κοινωνικό μοντέλο ως μια οντότητα οικονομική και νομική για να βελτιώσει την κατάσταση. Πρέπει να είναι πιο δυνατή η Ευρώπη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Όλε Σμιτ. ο Όλε Σμιτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σουηδική Προεδρία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συγχαρητηρίων. Ο Πισματάρης στην Πράγα τελικά υπέγραψε. Και ελπίζω ότι δεν θα μας απασχολήσει θεσμικά επί την επόμενη δεκαετία ο Βλάγκλαβ Χάβελ, πραγματικός ήρωας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν έτοιμο να κάνει κάποια βήματα σήμερα. Το ότι η τσεχική δημοκρατία απέκτησε τη δυνατότητα opt-out από τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι ατυχε, όπως είναι και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Κοπενχάγη αναμένεται συμφωνία όπου εκεί οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να υπομιστούν τις ευθύνες τους έναντι των φτωχών. Οι φτωχοί πλήττονται πιο σκληρά. Και τέλος, Υπουργέ, η διαδικασία προς τη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα όπου θα γίνουν οι διορισμοί είναι κάτι που έπρεπε να γίνει πολύ πιο ανεκτά διότι έτσι που γίνεται είναι ενοχλητικό για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, είναι ντροπιαστικό και δεν είμαι μόνο εγώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προβώ σε τρεις ε, παρατηρήσεις. Με τη συνθήκη της Λισαβόνα σε ισχύ χρειάζεται περισσότερο αποτελεσματική κοινή ε, εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική ασφαλείας που θα βασίζεται σε αλληλεγγύη. Μόνο τέτοια πολιτική θα εμποδίσει να επανεληφθούν άλλες πράξεις του Πούτιν. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι σε αυτή τη νέα κατάσταση να έχουμε συνεχώς μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να αναλάβει ευθύνες όσον αφορά την υλοποίηση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και τρίτον όσον αφορά τις υψηλές θέσεις τη καινούργια, χρειάζεται πρώτα απ' όλα θάρρος για να προχωρήσουμε και να υποστηρίξουμε όχι χαρτοφυλάκια αλλά προσωπικότητες. Προσωπικότητες που έχουν μακροπρόθεσμα οράματα και θέλουν να ε, συνεχίζουν και να προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Λοιπόν, αυτό για να αντιμετωπιστούν τεράστιες νέες προκλήσεις. Εκεί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικούς ηγέτες ευρωπαϊκούς όπω ε, τύπου Αντενάουρ, Σούμαν και θα πρέπει τις προσωπικότητες να επιδιώξουμε χωρίς προκαταλήψεις και θα πρέπει αυτοί οι ηγέτες ε, να βρεθούν και στα νέα κράτη-μέλη που σίγουρα θα πρέπει να εκπροσωπούνται στη μελλοντική Τρόικα. Ο Βάκλαβ Χάβελ σήμερα μας είπε ότι η Ευρώπη είναι η πατρίδα των πατρίδων μας. Και βάσει αυτού, αν το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε όσον αφορά την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ κύριε Κέλαμ. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Σάντρα Καλνιέτ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου διότι η συνθήκη της Λισαβόνας τελικά θα ισχύσει Πώς λοιπόν πρέπει τώρα να... Ε, ε, τι προσωπικότητα πρέπει να έχει ο πρόεδρος ε, που θα επιλεγεί. Θα πρέπει να μπορεί να παρακάθεται με τους αρχηγούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της αύριο και η ε, πρόεδρος της ε, ε, Λετωνίας Φράια Μπέργα είναι μια τέτοια πολιτική προσωπικότητα ηγετική η οποία θα μπορούσε να αναλάβει επιτυχώς αυτό το έργο η μοίρα της ε, ε, αντικατοπτρίζει ε, τη διηρημένη ήπειρό μας. Είχε φύγει από τη Λετωνία και επέστρεψε μετά την απελευθέρωση. Κατά τα 8 χρόνια της απουσίας της έγινε η Λετωνία μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρόκειται για μία προσωπικότητα η οποία θα φροντίσει τους πολίτες και θα μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό παρακαλώ, μην ξεπεράσετε το χρόνο κύριε συνάδελφοι, εσείς και οι επόμενοι ομιλητές. Ένα λεπτό κύριο Σταμπάτσι. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, κυρία Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας καταρχήν κυρώθηκε από την Ουγγαρία και θα ήθελα να συγχαρώ εν ονόματι όλων των Ούγγρων την, ε, την Προεδρία της Σουηδίας για την εξαιρετική εργασία. Βρήκαμε έναν φίλο των Τσέχων στο πρόσωπο της ε, Σουηδίας και μπορέσαμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ε, Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω καταρχήν ε, να ε, αντικατοπτρίσει η συνθήκη της Λισαβόνα στα δικαιώματα των πολιτών και θα ήθελα η κυρία Βάλστρομ να μας εγγυηθεί ότι οι επόμενοι επίτροποι θα εγγυηθούν τα δικαιώματα των προσφύγων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Ιρλανδία μας ρωτούν. Είναι ανυπόμονοι τώρα που επικυρώθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας. Με ρωτούν, είσαστε ανυπόμονοι, όχι γιατί χρειάστηκε τόσο απαντώ και κράτηση η γέννα τόσο πολύ. Ναι, υπάρχει ανακούφιση μεν και κάποια χαρά, αλλά βλέπουμε όπως και συζήτησε ότι τώρα ξεκινάει πραγματική δουλειά. Και είναι δύσκολη δουλειά να διοριστούν οι σωστοί άνθρωποι. Δεν είναι κάτι για παιδιά αυτές οι θέσεις, αλλά θέλουμε σε πολύ σημαντικές θέσεις να μπουν πολύ σωστοί άνθρωποι. Λυπούμε που χρειάζεται κι άλλος χρόνος για να γίνει αυτό διότι ε, καθυστερεί η τελική διαμόρφωση όλων των θεσμών και έχουμε πολλή δουλειά. Ίσως καλύτερη αυτή η καθυστέρηση και να κάνουμε σωστά τη δουλειά και να μπουν σωστοί άνθρωποι στις θέσεις. Και αυτές οι ανώτατες θέσεις είναι σημαντικές και θα πετήσουν ανθρώπους ε, με αφοσίωση που θέλουν να βελτιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι απλώς να έχουν μια δουλειά και μια θέση. Και να πω τελικά, έχει δίκιο και ο Σμπαρόσο για του θεσμού. Πρέπει να εισακουστεί το κοινοβούλιο. Ακούστε προσεκτικά. Εμεί είμαστε πιο κοντά στο εκλογικό σώμα και άμεσα εκλεγόμεθα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λούχαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ τα όσα είπε ο πρόεδρος Άνφελτ και τον Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, υπήρξε κοινή θέση για τη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Η Ρουμανία έκανε ήδη βήματα για την καταπαλέμηση της κλιματικής αλλαγής και να μειωθεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Δεν αρκούν όμως αυτά τα μέτρα για να πετύχουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερο στόχο από τη μείωση κατά 20%. Θα πρέπει να τηρήσουμε κάποιες, να θέσουμε κάποιους όρους σωστούς για τη σωστή προσπάθεια. Θα πρέπει η μελλοντική συνθήκη να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και να, να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους μειώσεως εκπομπών από τις ανεπτυγμένες χώρες, συγκρίσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να βοηθήσουμε τις ανεπτυγμένες χώρες. Αλλά έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα, εδώ, στην αίθουσα αυτή, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση και τα τρία θεσμικά όργανα εκπροσωπούνται από γυναίκες. Την κυρία Βάλστρομ, που εκπροσωπεί μάλλον έχουμε από τη Σουδική Προεδρία γυναίκα την κυρία Βάλστρομ από πλευρά τη Επιτροπή και έχουμε και πρόεδρο, προεδρεύουσα του σώματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και θα ήθελα αυτό να το βλέπουμε πιο συχνά και να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες. Ξέρω ότι και η κυρία Βόλης και η κυρία Βάλστρομ έχουν ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που να συμπεριλαμβάνει γυναίκες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επιστολή προς τον κύριο Μπαρόσο όπου ζητάνε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες, να υπάρχει μια ίση κατανομή μεταξύ των ε, φίλων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι ξέρουμε ότι και ο πρόεδρος Επιτροπής μας στηρίζει. Όμως παρόλα αυτά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε συχνά. Δεν μπορεί μόνο μέσω των αντρών να εκπροσωπούμεθα. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για την αναφορά σας. Ο κύριος Φάσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω ότι στηρίζω την θέση της Τσεχίας. Νομίζω ότι πήγαν έτσι και αλλιώς στο συνταγματικό δικαστήριο, έπρεπε να περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου, οπότε πιστεύω ότι υπεύθυνα συμπεριφέρθηκε ο πρόεδρος της Τσεχίας. Είναι κάποιος που δεν ήθελε να επικρατεί ε, έλλειψη βεβαιότητας και γι' αυτό και πευθύθηκε στο σταγματικό δικαστήριο. Οπότε καλά έκανε και περίμενε. Τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει να ισχύει σε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρέχουσες αποφάσεις των κυβερνήσεων που λήφθησαν για να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση δεν ήταν αρκετές. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να συντονιστούμε περισσότερο και να μην παίρνουμε ad hoc αποφάσεις οι οποίες τελικά αποδεικνύονται μη αποτελεσματικές προκειμένου να στηρίξουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να έχει πραγματικούς επαγγελματίες. Κυρία έχει το λόγο για ένα λεπτό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 Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένη ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη η οποία θα εδράζεται σε καλύτερη βάση και θα μπορέσει καλύτερα να επιλύει τα προβλήματα των πολιτών. Πρέπει όμως να ξέρουμε ποιο τίμημα πληρώσαμε διότι οι αξίες μας υποβαθμίσαν και ε, ο πραγματισμός υπερίσχυσε των αξιών μας. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρώπη ακολούθησε τις πιέσεις του Τσέχου Προέδρου και γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ ότι πάρα πολλοί ε, Ούγγροι και Γερμανοί ε, είχαν εκτοπιστεί δια της ε, βίας και έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτή ούτε πολιτικά ούτε ηθικά ούτε κοινωνικά. Όταν λοιπόν ε, συνδυάσουμε το έγγραφο αυτό με τις διαπραγματεύσεις ε, προσχωρήσεως μίας χώρας σαν την Κροατία το παράδειγμα είναι πολύ κακό και δεν θα έπρεπε να το, να το απορρίψουμε. λοιπόν που φτάσαμε εδώ. Η κυρία Τιτσάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καλωσορίζουμε την βαλτική στρατηγική, τη στρατηγική που διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή του Δούναβη αυτή η στρατηγική και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη και τέλος στη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι εξίσου σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει στη διάσκεψη της Κοπενχάγης ως ηγέτη στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η Ένωση ήδη μονομερός έχει θέση του στοχου 2020 20 Το πακέτο για την αλλαγή του κλίματο είναι ακόμα του κοινοτικού δικαίου και πρόκειται να εφαρμοστεί. Ζητώ η Ευρωπαϊκή Ένωση γρήγορα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο καινοτόμο και αποτελεσματικό για τη χρηματοδότηση οικονομία φιλική και οικολογική, φιλική προ το περιβάλλον και οικολογική. Θα πρέπει να χρηματοδοτούνται τα μέτρα τη Ένωση για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματο. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει επενδύσει στη βιομηχανία και στι δημόσιε υπηρεσίε, ώστε να δημιουργούνται θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Έχει για ένα λεπτό. Tehát elnök Ευχαριστώ. Κύριε Βάλστρομ. Έχουν περάσει ήδη 20 ε, χρόνια που έπεσε το σιδηρού παραπέτασμα ε, ε, στην πολιτική σκέψη ίσως δεν έχει καταργηθεί ακόμη και υπάρχουν ε, παλιά κόμπλεξ. Σκεφτείτε τις διαδηλώσεις ε, των, ε, στην Ουγγαρία πριν δύο χρόνια που καταπατήθηκε πολλοί κόσμος και υπάρχουν ακόμη παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μειονότητες δεν, έχουν, δεν χαίρουν των δικαιωμάτων τους ε, η ε, συνθήκη της Λισαβόνας περιγράφει ορισμένες αρμοδιότητες τις οποίες πρέπει να σεβαστούμε και όποιος επίτροπος αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει επίσης να σκέφτεται και τις μειονότητες, τις γλωσσικές μειονότητες που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή διότι ε, έχουμε εδώ υπευθύνου, οι οποίοι πρέπει να λύσουν τα προβλήματα και να στηρίξουν αυτούς που συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, η στήξη Αβώνας, τελικά έγινε αποδεκτή, επικυρώθηκε ενισχύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται αποτελεσματικότερη στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να υιοθετήσουμε ε, διάφορες αποφάσεις και όσον αφορά και τη συνεργασία μεταξύ των νέων ηγετών, των νέων καθηκόντων που θα πρέπει να αναλάβουν ε, οι νέες θέσεις της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει να κρυβούμε όμω και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η καταπολέμηση τη οικονομική κρίση είναι ένα στόχο άμεσο. Η καταπολέμηση τη ανεργία ή μια εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Κοπενχάγη είναι κάτι απαραίτητο και θεμελιώδε, αλλά σε αυτή τη φάση των κρίσεων δεν είναι η καλή στιγμή για να αποφασίσουμε ε, ποιε χώρε, ποιοι διεθνεί φορεί ε, θα δώσουν χρηματοδοτήσει και ποιε θα είναι οι υποχρεώσει που θα αναλάβουν. Η λύση των προβλημάτων των οικονομικών και των κοινωνικών σε αυτή τη φάση αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητα για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Σκέλη έχει το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή που μαζί με την κυρία Μαγκίνης είμαι εδώ στη δέκατη επέτειο από την πτώση του τείχους και παραμονές ε, της θέσεως ισχύ της ε, συνθήκης της Και πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερο προνόμιο ότι η Ιρλανδία ψήφισε με 67% υπέρ της συνθήκης της Λισαβόνας και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη έγκριση τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί σειρά ετών. Επίση, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμο θα δει την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τους εμφύλιους πολέμους που ακολούθησαν μετά σε πολλές χώρες, όπως και στη χώρα μου. Όταν ήρθε η ελευθερία στη χώρα, οδήγησε εμφύλιο πόλεμο. Και εκεί βλέπουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έδινε προσανατολισμό και υποστήριζε τις χώρες εκείνες. Και τελικά δεν δόθηκαν οι εμφύλοι πόλεμοι λόγω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα μιλάμε για το ποιοι θα καλύψουν τι θέσει αυτέ που δημιουργήθηκαν. Το είπατε εκπροσώπου και του πρόεδρου. Αν ο πρόεδρο δεν είναι πρόεδρο για να είναι πρόεδρο και είναι. Να το πούμε πρόεδρο με την έννοια του πρόεδρου μια επιτροπή, όχι πρόεδρο με την έννοια ενό πρόεδρου τη Δημοκρατία. Ο κύριο Μίτσελ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, χάρηκα πάρα πολύ που στη Στοκχόλμη ε, στα πλαίσια των ημερίδων ανάπτυξη, επισκέφθηκα του χώρου όπου οργανώθηκαν διάφορε εκδηλώσει και συμμετείχα και στην ε, συζήτηση που έγινε στο Ιρλανδικό ραδιόφωνο για τι Υπηρεσίε. Κάποιο έλεγε ότι μειώνουμε τι δαπάνε για την υγεία ε, για την ανάπτυξη και εγώ έπρεπε να εξηγήσω ότι το θέμα δεν είναι ότι αν κόψουμε από το ένα μπορούμε να δώσουμε στο άλλο, όχι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, και για την υγεία και για την ανάπτυξη. Οπότε λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την ανάκαμψη στην Ευρώπη, πώς αντιμετωπίζεται η κρίση οικονομική στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή μην ξεχνάμε ότι 11 εκατομμύρια παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο πεθαίνουν καθημερινά πολλά από αυτά γιατί δεν έχουν φάρμακα, το οποίο εμείς είχαμε 30 χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το έχετε αυτό υπόψη σας, να υπάρχει στην ατζέντα πάντα. Και όταν κάποιος οριστεί για τις εξωτερικές σχέσεις, μην ξεχνάμε ότι ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ριβελίνη έχει το λόγο. Mr. Ριβελίνη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου ε, λαμβάνουν χώρα 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Η πτώση του τείχους ήταν η απαρχή της πραγματικής Ευρώπης. 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια κατέρευσε ένας τείχος, ένα τείχος ε, που ήταν γεμάτος προκαταλήψεις, τυραννία, πείνα για πάρα πολλούς πολίτες της Ανατολής. Και σήμερα δεν πρέπει να γιορτάζουμε πλέον την πτώση του τείχους, αλλά θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι να κάνουμε μετά αυτό το τείχος. Διότι εν τω μεταξύ ψώθηκαν άλλα τείχη. Τα τείχη που χωρίζουν τι βόρειε με τι νότιε χώρε του πλανήτη, ε, οι πιο ανεπτυγμένε χώρε και οι πιο φτωχέ, χώρε που παράγουν προϊόντα και χώρε που παράγουν ιδέε. Πιο ψηλά τείχη και πιο δύσκολα να καταρρεύσουν και μπορεί σε όλη την ανθρωπότητα να δημιουργήσουν ε, μεγάλε δυσκολίε και πολέμου. Γι' αυτό ο διορισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά τη Λισαβόνα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτοί οι διορισμοί δεν μπορούν να γίνουν με απλώς διορισμό κάποιων μέσα σε μυστικές συνεδριάσεις. Χρειάζεται να υπάρχει μια συνεισφορά ε, να, θα πρέπει να συμβάλλει όλη η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συμβάλλουμε, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν ε, γκρεμίσουμε αυτό το τείχος του nomination, του διορισμού, που επιλέγει τους μελλοντικού υποψηφίους μέσω ισορροπιών μεταξύ χωρών και όχι μέσω προσόντων, τότε θα έχουμε κάνει την Ευρώπη των Εθνών. Ευχαριστώ. Αλλά πολύ το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Ε, τώρα, τελευταία παρέμφαση, ε, τον κύριο Μπρόνς. Mr. Andrew Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ηγέτης αντιπολιτεύσεως της Βρετανίας δήλωσε ότι θέλει να επαναδιαπραγματευτεί κάποια τμήματα συνθήκης της Λισαβόνας αυτό χρειάζεται όμω ε, και τη συνένεση και των 27 κρατών μέλων. Ανακοίνωσε και την εισαγωγή ενό νόμου για την κυριαρχία που θα υποχρεώσει η διεξαγωγή δημοψηφίσματος εν ώψη νέων συνθήκων. Αυτό μπορεί ε, να απορριφθεί από επόμενε κυβερνήσει, να αποσυρθεί. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν ότι οι συντηρητικοί ηγέτε, τα σχέδια του συντηρητικού ηγέτη είναι πομφόλιγες και το κόμμα το αποφάσει ή θα αποφασίσει να δεχτεί τη συνθήκη τη αγώνα ή ακόμα καλύτερα να βγάλει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελείωσαν οι παρεμβάσει των βουλευτών και το λόγο θα πάρει η κυρία Μάλστρομ εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια. Η Σουηδική Προεδρία συμμερίζεται τη χαρά σα για το γεγονό ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα επιτέλου έχει επικυρωθεί από όλε τι χώρε. Αυτό μα δίνει μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική και μα επιτρέπει να έχουμε ένα πιο ενισχυμένο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Συμφωνώ επίσης με εκείνου από εσά που είπαν ότι ίσως είναι σύμπτωση, αλλά πάντως είναι μια εβδομάδα που πολύ καλά διάλεξε ο πρόεδρος Κλάους για να υπογράψει την συνθήκη. Αυτή τη βδομάδα που έχουμε και την επέτειο από την πτώση του σδηρού περαπετάσματο, την πτώση του κομμουνισμού και την αρχή της Ευρωπαϊκής ενότητα και την τελική νίκη των ιδεών του Σούμαν και όχι του Στάλιν. Και τώρα μια που μιλάμε για την Τσεχία. Θέλω να επιβεβαιώσω για τον κύριο Νταφ ότι οι Τσέχοι δεν πήραν γενικό opt-out για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι. Υπάρχει πάντα η συνθήκη που ισχύει, αλλά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για ορισμένες χώρες, όπως η Αγγλία κλπ, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι η Επιτροπή και το Δικαστήριο που θα κάθε φορά εφόσον υπάρξει ε, μια δυσκολία. Τώρα, όπω είπε και ο πριν φύγει, οι διαβουλεύσεις με τους 26 συναδέρφους συνεχίζονται. Η δουλειά είναι σκληρή. Φιλοδοξεί, αισιοδοξεί την επόμενη πέμπτη να έχει κάτι παραπάνω. Βέβαια είναι πολύ πρόημο να μιλάμε για ονόματα. Και εγώ διαβάζω τις εφημερίδες και εγώ έχω ακούσει ονόματα, ονόματα που δεν θέλετε, ονόματα που θέλετε. Ναι, άκουσα και από εσά για κανένα δύο. Εντάξει, ό,τι υποψηφιότητε έχετε και δικέ σα ευχαρίστω να τι δώσετε στον πρόεδρο, θα τι μελετήσουμε. Υπάρχει περιθώριο μέχρι την Πέμπτη. Και βέβαια, ακούμε όλες σας τις ανησυχίες για να υπάρχει ισορροπία περιφερειακή μεταξύ των δύο φύλων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πιστεύω και εγώ αυτό, πρέπει να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι την Ευρώπη δεν τη διαχειρίζονται μόνο οι άντρες. Αλλά δύο θέσεις ε, έχουμε να μοιράσουμε και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλες οι προϋποθέσεις να καλυφθούν. Είναι δύσκολο, αλλά ακούμε. Ό,τι συμβουλές έχετε, ό,τι ανησυχίες έχετε, τις ακούμε. Τώρα, για τον είπα το εκπρόσωπο. Αυτός ή αυτή θα ολοκληρώσει το πλαίσιο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τις εξωτερικές σχέσεις. Και αυτό από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν υποβληθεί στο Συμβούλιο το αργότερο τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Όπως πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε πει, ο ύπατος, η ύπατος εκπρόσωπος θα παρακολουθεί τις συζητήσεις και θα απαντάει στις ερωτήσεις σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αληθούν οι απόψεις σας στην ε, πολιτική που εκπονούμε. Τώρα στην Μελίτα Όσκουρτ που νομίζω έφυγε, θέλω να πω ότι η Συνδική Προεδρία δεν έχει παραιτηθεί καθόλου από τις φιλοδοξίες της για τις διάφορες στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Κάθε άλλο. Θέλουμε τις φιλοδοξίες μας ε, να τις κρατήσουμε. Ίσως όχι τώρα αμέσω, αλλά πολύ σύντομα. Αν αφήσουμε τις οικονομίες μας να συνεχίζουν να δημιουργούν ελλείμματα, καταλαβαίνετε ότι οι πιο ευάλωτοι στις κοινωνίες μας θα την πληρώσουν. Δεν το θέλουμε αυτό. Βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Σίγουρα πολλές χώρες υποφέρουν από υψηλή ανεργία και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε αμέσω την ε, στρατηγική εξόδο από την κρίση. Αλλά υπάρχει σαν σχέδιο και θα γίνει αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία να περάσουμε στι επόμενε γενιές. Τέλο, για το κλίμα κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν έχουμε μειώσει τι φιλοδοξίε μα. Η Συνδική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και πολλοί άλλοι δουλεύουμε μέρα νύχτα. Είμαστε πεπισμένοι για τι θέσει μα δουλεύουμε σκληρά και έχουμε διαπραγματεύσεις για να προχωρήσουμε. Πάρα πολλές συναντήσεις και πάρα πολλές ακόμα θα γίνουν, ακόμα και αν μένουν μόνο 25 μέρες μέχρι την Κοπεχάγη. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ε, ανησυχεί και το βλέπω αυτό. Και είναι πολύ αθαρρυντικό ότι ο κόσμος ζητάει λύσεις, αλλά δεν φτάνει αν θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο των δύο βαθμών δεν υπάρχουν όλα τα κομμάτια του παζλ έτοιμα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία. Είναι ένα γεγονός, δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά έτσι είναι. Συνεχίζουμε να το προσπαθούμε, αλλά δεν θα γίνει, γιατί πολλές πλευρές λένε ότι δεν είναι έτοιμες να κάνουν αυτό το βήμα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ηγετικό ρόλο και εξακολουθούμε να δουλεύουμε για μια φιλόδοξη συμφωνία με ένα πλαίσιο όπου να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εταίροι και ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο στόχος μας είναι ε, το Κιώτο να προχωρήσει με δεσμευτική συμφωνία. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την δουλειά του. Ξέρω ότι κάνετε πολλά και θα συνεχίσουμε και μετά την Κοπεχάγη. Η Ευρώπη έχει ακόμα ηγετικό ρόλο εξακολουθούμε, έχουμε τις υψηλότερες φιλοδοξίες μέχρι τώρα, το έχουμε επιβεβαιώσει και τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις στηρίζουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το ρόλο μας. Θα είμαστε ένα στοιχείο κλειδί προκειμένου να ε, πετύχουμε τους στόχους μας, να υπάρξει σωστή κατανομή του βάρους, αλλά σας είπα μερικές πλευρές δεν είναι έτοιμες και δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς νούμερα. Θέλουμε να πιέσουμε, αλλά και ξέρουμε ότι και άλλοι πρέπει να πληρώσουν, είναι προς το συμφέρον όλων. Σας ευχαριστώ πάντως για την ενθάρρυνσή σας και προσδοκούμε να συνεχίσουμε τις συνεργασίες μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Μίλησε γαλλικά η Σουηδή υπουργό, θα πρέπει και εγώ να μιλήσω σουηδικά λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Προέδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να μιλήσω σουηδικά και να πω κάποια πράγματα για κάτι σημαντικό που εθίγει σήμερα. Δηλαδή, πως το κείμενο της νέας συνθήκης μπορεί να ενταχθεί στην πραγματικότητα την οποία θέλουμε να αλλάξουμε. Πώς το κείμενο της νέας συνθήκης της Λισαβόνας μπορεί να μας δώσει κατεύθυνση, προσανατολισμό και τα εργαλεία για να πάρουμε τις αποφάσεις σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, και όσα ακολουθούν κοινωνικά προβλήματα, ανεργία, πώς θα αντιμετωπίσουμε μεταναστευτικά προβλήματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε άλλες πτυχές που έχουν προτεραιότητα, πώς συσχετίζονται όλα αυτά, όπως ανέφερε και ο κύριος Μπαρνιέ νωρίτερα σήμερα. Αυτό βέβαια αφορά και την εφαρμογή, την εκτέλεση. Ποιους θα διορίσουμε ε, ως εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως ποιος θα είναι ηγέτης, ποιοι θα είναι ηγέτες στις υψηλές θέσεις, ποιοι θα διοριστούν εκεί. Και όπως θα γνωρίζετε, ο σωστός άνθρωπος, η σωστή δουλειά, πολύ συχνά είναι γυναίκα. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ. Ευτυχώς γνωρίζω ότι έχω και πίσω μου τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ακολουθείται μια δημοκρατική διαδικασία και αυτό είναι σημαντικό. Η διαδικασία που ξεκίνησε είναι δημοκρατική και παρέχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δείξουν ότι δεν είναι θέμα απλώς να λένε λόγια, αλλά ότι θα πρέπει να επιλεγούν έξυπνοι, ε, αρμόδιοι υποψήφοι, υποψήφιες γυναίκες που μπορεί να προωθηθούν. Διαφορετικά εμείς που είμαστε η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εμείς η πλειοψηφία είμαστε οι γυναίκες, θα πρέπει να μπορούμε να πάρουμε και τις δημοκρατικές αποφάσεις. Αυτό που είπε ο Βάκλαφ Χάβελ. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό και δεν είναι κάτι αμετάκλητο. Η δημοκρατία πρέπει να θρέφεται, πρέπει να τρέφεται και πρέπει να πολεμούμε για δημοκρατία και ξανά και ξανά και ξανά, πανηλημμένα. Ε, συνεργαστήκαμε στενά με τη Σουηδική Προεδρία για μία ακόμη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την σκληρή δουλειά που έκαναν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρου μου, θα του ευχαριστήσω και για τη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια απόφαση σήμερα, όπω είπε και ο κύριο Μπαρόσο. Πήρε απόφαση λοιπόν σχετικά με το πρώτο μέτρο για το οποίο πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη. Την πρωτοβουλία για τους πολίτες όπως αποκαλείται ξεκινήσαμε ε, διαδικασία διαβούλευσης, μια πράσινη βίβλο που περιέχει 10 ε, ερωτήσεις. Και αν πάρουμε καλές απαντήσεις μέχρι ε, τέλος Ιανουαρίου, τότε ελπίζουμε η διαδικασία να είναι ταχεία μέσα του Κοινοβουλίου και αυτή η πρωτοβουλία για τους πολίτες, για την Ιθαγένεια, να μπορεί να προωθηθεί και να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του επομένου έτους. Αυτό θα δείξει άριστα το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες ρήτρες, τις νέες διατάξεις, τις νέες δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνα για να δώσουμε στους πολίτες μεγαλύτερη επιρροή και περισσότερο λόγο. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα ήδη σχολιάστηκαν από πάρα πολλούς αγορητές και από την Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε είναι να μιλάμε με μία φωνή ε, συνεχίζοντας να επιμένουμε ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι ισχυρή και δεσμευτική βεβαίως ε, το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία είναι κάτι που θα εξετάσουμε αφού δούμε τι έχουν να πούν και οι εταίροι μας ποιες θα είναι οι διαπραγματευτικές τους θέσεις οι προσφορές και αντιπροσφορές τους και τέλο, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα, τη στενή συνεργασία μας όσον αφορά την εκτέλεση, την υλοποίηση της συνθήκη τη Αβώνα. και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που, να, που μπορώ να διαβιβάσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη απόψη του Κοινοβουλίου. Εμεί είμαστε θεματοφύλακες ε, των συνθήκων και βεβαίω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι εμείς θα τηρούμε τη συνθήκη κατά γράμμα. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Vice President. Η συζήτηση σέλιξε εδώ. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιάς μας διάταξης που προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας της 18ης Νοεμβρίου του 2009 στη Στοκχόλμη. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την ε,